Welcome to this meeting. Καλώς ήρθατε. Το σχέδιο ημέρησης διάταξης ελπίζω ότι μπορεί να εγκριθεί με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Η ψηφοφορία για το σημείο 5, επισφαλή συμβόλαια εργασίας, δεν θα εξεταστεί σήμερα, έχει αναβληθεί. Και όπως ξέρετε, Έχουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα για τη συνεδρίασή μας. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε το απόγευμα στις 2 και όχι στις 3. Έχουμε μια πιο σύντομη διακοπή μεσημεριανή, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να τελειώσουμε τη συνεδρίαση εγκαίρως για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο ή στον σταθμό του τρένου. για τους διερμηνείς επίσης. Θα επιστρέψουμε στις 2 η ώρα. Όλες οι γλώσσες είναι, είναι διαθέσιμες εκτός από τα μαλτέζικα και τα κροατικά. Έχουμε 17 ε, επισκέπτες οι οποίοι θα κάψουν και θα μας ακούσουν. Τους κάλεσε η κυρία Αέγνα η οποία θα έρθει σε λίγα λεπτά. Ναι, έχουμε και μαλτέζικα. Όλο εξαιρετικά. Αν τα θέλετε βέβαια, αν δεν τα θέλετε δεν τα έχουμε. Έγκριση των πρακτικών της 1ης Απριλίου και της 16ης Απριλίου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα έχουμε εγκρίνει. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Και ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Έχετε την κάρτα σας ψηφοφορίας. που θα ξεκινήσουμε με το κείμενο συμβιβασμού που έχει εγκριθεί από την ε, Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων επί της προτάσεως της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ναυτιλωμένους. Τελικός ε, κατάλογος προφορίας για την συμφωνία με το Συμβούλιο ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. «42 προς 1 με καμία αποχή». Συγχαρητήρια. Και σας ευχαριστώ τα μάλλον. ή την κυρία Μωράν Σατιέ ιδιαίτερα που ήταν και η αρμόδια για το θέμα αυτό. Πάμε τώρα στο σημείο 6, γιατί το 5 έχει αναβληθεί. Τροπολογία 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 123 έχει αποσυρθεί. 19 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά δεκτή τροπολογία 23 υπέρ κατά δεκτή 126 ψήφι υπέρ κατά δεκτή Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 126, έρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. Συμβαστική KA ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 128, 129 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 129. Αρχιέται η ψηφοφορία. Πέρασε δεκτή. 26-23. Συμβαστική L υπέρ. Συμβαστική M υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος. Βεβαίως. Για την 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ιδίας αυτής ψηφοφορίας εγκρίνεται. 100 <coughs> τροπολογία 30 μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1.35 υπέρ. Α, εκπίπτει. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25, καθώς και 140 και 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική N <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ιδίας. Εγκρίνεται. 77 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Okay. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 όχι εκπίπτει. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή οι δύο εκπίπτει τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία συγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές δεκτή. 99 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 103. Ανοίγει η ψηφοφορία. Πέρας. Ενεκρίθη πράγματι. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 104 άρχεται πέρασε, απορρίπτεται 105 υπέρ κατά άποχες απορρίζεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 και 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 38 με 10 και 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κύριο Λένας. item 7. Περνάμε στο σημείο 7 για την έρευνα και την καινοτομία για τη δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη. Αρχίζουμε με τη συμβιβαστική A, υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9, συγγνώμη, τροπολογία 9, υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Αν θέλετε έλεγχο. Όχι, όχι, ήταν πολύ σαφές. Καλά. Ας την ελέγξουμε την 9. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίψετε. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 με προφορική τρομολογία από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Για περισσότερα αξιόπιστα δεδομένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος τη 16. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ κατά εποχές να την ελέγξουμε. Την τροπολογία 28 έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 34 Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Έναρξη της ψηφοφοριας περας Πέρασε. Εγκρίνεται 27-23. Τροπολογία 35 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική DA, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε τη τροπολογία 44, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους. Διαφορά. 45. Υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα δεύτερο τμήμα υπήρχε που πρέπει να το ψηφίσουμε. Είναι προσθήκη στη συμβιβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε την τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. And it's carried by 51. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο σημείο 8. Σχέδιο δρομηγότηση τη κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε για την εφαρμογή τη αρχή των ίσων ευκαιριών και τη ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία και την αποσχόληση. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος της 17 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έξι ψήφι διαφορά. 18. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος Τις 18. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική B. Υπέρ. <coughs> Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Με προφορική τροπολογία από τους πράσινους. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Με προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε την 26. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Μία ψήφος διαφορά. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. αποχεύ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική E υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος τη συμβιβαστική G έναρξη ψηφοφορίας πέρασε Εγκρίνεται. 12 ψήφοι διαφορά. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε την τροπολογία τέσσερα. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο τη γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε, έναρκη, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 42-8. Yeah. we vote on uh, the draft opinion by Madam Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Μάκιντάι για το πρόγραμμα ReFit, τροπολογία υπαριθμών 1 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία υπερτιμών 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Με τρεις ψήφους ε, υπερ, Συμβαστική α. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική ΑΑ καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν μπορούμε συνεχώ να επαναλαμβάνουμε με ηλεκτρονική επαλήθεια. Συμβαστική ΑΑ ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και γκρίνεται. Η 15 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 14 καταπίπτει. Η 13 ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 15 τώρα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Γιατί 15. Τροπολογία υπαριθμών 15. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για τη 15. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο ε, υπέρ. Μία ψήφο διαφορά. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Για την 12. Ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 12. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάλι με μία ψήφο διαφορά. Η 16. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 17. Όχι. Ψηφίζουμε για τη 17 μάλιστα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. Η συμβιβαστική Β ηλεκτρονικά Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Απορρίφθηκε, ναι, ναι, έχετε δίκιο, απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 20 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε και για την 18. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε τώρα η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Η 21 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. 27 παρακαλώ ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Η 28 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία και γκρίνεται. Η 29. Το πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε παρακαλώ. η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε για το τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Η 30. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 31. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική A Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική M. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 44. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Συμβιβαστική K. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία 46. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Για το πρώτο τμήμα τη 46 ψηφίζουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Η 48. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 48. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Η 49 η 51, 52, 53 και ψηφίζουμε παρακαλώ. Και τώρα έκλεισε η ψηφοφορία, απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Ψηφίζουμε για την 54. Καταρχήν δεν κατάλαβα. Γιατί ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε γιατί τελικά μου δεν είναι και σπουδαία. Ερωτώ. Γιατί ψηφίζουμε για κάθε τροπολογία ηλεκτρονικά. Γιατί εξοικονομούμε χρόνο, λέει η πρόεδρο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία για την τροπολογία υπερθυμών 54. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 55 ψηφίζουμε. Ξεκολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. 59 τώρα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 56 καταπίπτει. 70. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε τώρα η ψηφοφορία και εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Η 69, όχι καταπίπτει η 69. Για την 74 ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Και εγκρίνεται η τροπολογία υπαριθμών 74. 75. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. κλείσει η ψηφοφορία και εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 76. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Εγκρίνεται 77. Λοιπόν, Ψηφίζουμε τώρα για την 77. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 78. Με προφορική τροπολογία ψηφίζουμε παρακαλώ. Τώρα έκλεισε η ψηφοφορία. <clears throat> Απορρίπτεται. Η 79. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Η 80. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική ε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Και απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 81. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 85 καταπίπτει η 94 της κυρίας Χάρφκιν ψηφίστε παρακαλώ έκλεισε ψηφοφορία και γκρίνεται 96. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο. 97 ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται 98 ψηφίζουμε. Και έκλεισε τώρα η ψηφοφορία και απορρίπτεται με μία ψήφο συμβαστική F. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. την 110. 11 και 12. Ψηφίζουμε για τις 3. 110 και 112. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. Καταπίπτει. Η 121. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Πρέπει να πάμε πίσω στην 120. Ψηφίζουμε για την 120 παρακαλώ. Ψηφίσαμε τώρα, έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. ψηφίζουμε για την 123. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 123, 124, 125 και 126 από κοινού και γκρίνονται αυτές οι τροπολογίες. Πάμε στην H, στο, ε, στην τροπολογία H. Αλλά αυτή καταπίπτει. στην ΆΗ. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την ΆΗ, τροπολογία ΆΗ. Έκλεισε ψηφοφορία και εγκρίνεται η τροπολογία. Πάμε στην 137 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική L. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 140 Ψηφίζουμε για την 140. Κλείνει, έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. 141 μαζί με την 122 παρακαλώ ψηφίζουμε για αυτές τις δύο. Πάμε στην ε, ναι, για την 122 ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Για την 144 ψηφίζουμε. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Συμβιβαστική J Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 145. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Μισό λεπτό. Τώρα έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 151 ψηφίζουμε. Τροπολογία 152. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η 155 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 156 ψηφίζουμε γιατί είναι 156 εγκρίνεται 157 ψηφίζουμε παρακαλώ. Τώρα έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται. 158 καταπίπτει, πάμε στην 159. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 160 πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται, πάμε στο δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. 161. Ψηφίζουμε για την 161 παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίφθηκε και ψηφίζουμε κατόπιν τούτου για το σύνολο της ε, ε, γνω, τροποποιημένης γνωμοδότησης, σχεδίου γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Ξανά, από την αρχή. Από την αρχή λοιπόν ε, ψηφίζουμε ονομαστικά για το σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Τώρα ψηφίσαμε όλοι, άρα κλείνει η ψηφοφορία και εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότησης. Καλώ, λέει η Πρόεδρος. Διαφημιστικό διάλειμμα. Yeah.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 Okay, friends, thank you for... Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Τώρα, να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Τομπρόφσκης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τον γνωρίζουμε όλοι. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ σήμερα και είναι εδώ επίσης και η Επίτροπός μας, η κυρία Τάισεν, τώρα μια ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με τον κύριο Ντομπρόφσκι και την κυρία Τάισεν. Όπως πάντα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί όταν θέτουμε τα ερωτήματά μας και εκφράζουμε την άποψή μας κατά τη συζήτησή μας, να αρχίσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκι για την παρουσίασή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου και που έχω τη δυνατότητα να έχω μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας σε σχέση με την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα αποτελέσματα μετά από 7 μήνες από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπα σε, στην ακρόαση τον προηγούμενο Οκτώβριο ότι ο ρόλος μου ως Αντιπροέδρου ε, είναι ακριβώς ε, τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα να ε, θεωρούνται ίσα και να ενισχύσουμε βεβαίως τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξή σας όσον αφορά ε, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ε, ατζέντα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα καταρχάς να πω ορισμένα πράγματα για την πρόοδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ειδικότερα σε σχέση με τις πρόσφατες συστάσεις αναχώρα, όπως ε, και την εφαρμογή του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επίσης, η Επίτροπος Τάισεν θα μας κάνει μια πιο λεπτομερή παρουσίαση των τρεχουσών πρωτοβουλειών και των ε, σχετικών εργασιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλουμε να αυξήσουμε την ε, ε, κυριότητα ε, και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, ειδικότερα με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων και Εθνικών Εταίρων. Ο ενισχυμένος ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικότερος από ποτέ για να ενισχύσουμε αυτή την αίσθηση της κυριότητας και της λογοδοσίας. Το, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2015 ε, το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής. Είναι το επίκεντρο της ολοκληρωμένης μας προσέγγισης η οποία επικεντρώνεται στις επενδύσεις ε, και στην δημοσιονομική ευθύνη. Αυτό βέβαια είχε άμεση σχέση με την ετήσια έρευνα ε, για την ανάπτυξη, νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις οποίες ε, θα υποβάλλεται και γνωμοδότηση, κάτι το οποίο φάνηκε σε εκθέσεις αναχώρα που δημοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο. Οι ειδικέ αναχώρα συστάσεις δημοσιεύτηκαν πριν από δύο εβδομάδες και αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο, στην ανάκαμψη που πρέπει να γίνει πιο σταθερή και πιο βιώσιμη. Τα μηνύματα είναι σαφή, πρέπει να υπάρξουν ε, πολύ μεγαλύτερες προόδου, ως προς το ε, τομέα του, της, του, της αγοράς εργασίας μεταξύ άλλων ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ενίσχυση της, της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης δείχνουμε τις προκλήσεις που είναι συγκεκριμένες για την κάθε χώρα και θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Πολλές από τις συστάσεις επικεντρώνονται στις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι πολύ σημαντικές για τις χώρες που έχουν κάποια καθυστέρηση ε, λόγω της κρίσης και πρέπει να επανέλθουν στο επιθυμητό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ε, ευκαιρίες απασχόλησης, να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα για τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία. Επίσης, ε, Υπάρχουν τομείς που καλύπτονται από τις προτάσεις μας ε, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας μας, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί σε απτά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι θα γίνει μια συνεδρίασή σας συγκεκριμένα στις 23 ε, Ιουνίου για τις ε, αναχώρα συστάσεις. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει τη διαφορά σε, στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, την αντικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτή η νέα αρχή για την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται στην, ε, στο εστιασμένο πρόγραμμα ε, εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι οι, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να διατηρήσουν την κεκτημένη ταχύτητα και τη δυναμική. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να προωθήσουμε ε, τη δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες. πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν στους πολίτες τους να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, να υποστηρίξουν την μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία για τους νέους, όπως επίσης και την κοινωνική συνοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερως που η πρόταση της 4ης Φεβρουαρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίσπευση της πρωτοβουλίας για την εργασία των νέων εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα παρουσιάσουμε περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση της, της απασχολησιμότητας σε μεταγενέστερο στάδιο φέτος και η Επίτροπος Τάισεν θα μας πει λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα στη συνέχεια. Να τονίσω επίση το εξή. Δύο σημαντικού τομεί ε, του προγράμματο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει να κάνει βέβαια και με τη δική σα εργασία. Η η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή ενισχύθηκε ιδιαίτερα ε, σε ε, προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Βέβαια, ε, χρειάζονται και άλλα βήματα για να υπάρξει σταθερότητα και για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανάγκες δημιουργίας θέσης απασχόλησης θα πρέπει να, να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα ε, στο πλαίσιο της διακυβέρνησης Ευρωζώνης ε, και θα γίνει ε, παρουσίαση σχετικής έκθεσης τον επόμενο μήνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης ε, θέλουμε ε, να αποτελέσει το επίκεντρο μιας το κοινωνικό ζήτημα να αποτελέσει το επίκεντρο μιας καλύτερης οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Μια, ένα πακέτο δύο, ένα, μια δέσμη δύο πακέτων μετά από την έκθεση αυτή που θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα, ε, θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ποια θα είναι ε, η συνέχεια όλης αυτής της προσπάθειας και ε, θα ενταχθεί και στο θεματολόγιο για την καλύτερη διακυβέρνηση. Αυτό βέβαια, ένα, μια, ένας καλύτερος συντονισμός του κύκλου πολιτικών θα έχει ως αποτέλεσμα μια νέα εστίαση στη διαβούλευση για την μεταρρύθμιση της διαδικασίας καθορισμού των πολιτικών. Ο κοινωνικός διάλογος τώρα. Ο κοινωνικός διάλογος ε, έχει ενισχυθεί, είναι ε, βασικό ε, επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προγράμματος Εργασίας. Έγινε ένα, μια, ένας διάλογος υψηλού επίπεδου και χαρήκαμε όλος ιδιαιτέρους που ο πρόεδρος Σούλτς ήταν εκεί για να χαιρετήσει τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων. Να σα δώσω ένα παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αυτό είναι ένα, ακόμη ε, μια, μια καλύτερη ένδειξη τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. όπω ε, είπα και προηγουμένω όταν ε, παρουσίασα τις προτεραιότητες της εργασίας, της εργασίας μας κατά την ακρόαση μετά τη δημοσίευση των, ε, των εκθέσεων αναχώρα ε, αναφερθήκαμε, παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία με τα εθνικά κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις, ε, τα κράτη-μέλη πριν από τις αναχώρα συστάσεις και θα συνεχίσουμε αυτές τις διαβουλεύσεις. Συζητούμε τώρα την εφαρμογή των εκθέσεων των ειδικών αναχώρα, όπως επίσης και την εστίαση ε, στις ε, ε, σχετικές πολιτικές. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια, με διάφορους εθνικούς φορείς για να μπορέσω να συζητήσω τέτοιου ή τις εκθέσεις αναχώρα και ειδικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εκθέσεις αυτές και σήμερα ε, θα πάω στην Κροατία στο πλαίσιο επίσκεψης, ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να συζητήσουμε τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην Κροατία την, αναχώ τη συγκεκριμένη ε, χώρα, τη συγκεκριμένη έκθεση αναχώρα. Ε, όσον αφορά τώρα τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι στην προσπάθεια ε, δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να, να ε, συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην απασχολησιμότητα και στο πακέτο κινητικότητας. Πέραν τώρα του χαρτοφυλακίου μου και στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για το πρόγραμμα εργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην Ενεργειακή Ένωση, στην ψηφιακή αγορά, στην ε, πολιτική ε, μετανάστευση, μεταξύ άλλων. Και πέρα από το πρόγραμμα ε, για το 2015, έχουμε προβεί σε ένα συλλογισμό για ένα στρατηγικό όραμα όσον αφορά ε, την κοινωνική πολιτική συγκεκριμένα. Ε, έχουμε συγκεκριμένη συνεδρία στις 9 Ιουνίου και η Επίτροπος Τάισεν θα πει περισσότερα όσον αφορά την πολιτική απασχόληση και την κοινωνική πολιτική κατά τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με χαρά θα ακούσω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης. θα δώσω το λόγο στην κυρία Τάισεν τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ενώπιον σας και πάλι. Θα ήθελα να προσπαθήσω να συμπληρώσω την εισαγωγή που έκανε ο Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόφσκη, αναφερόμενη πρώτα στην ακρόαση που κάνατε όταν ήμουν υποψήφια για επίτροπο τον προηγούμενο Οκτώβριο και επίσης σε συνάρτηση με τις προτάσεις που έχει εντοπίσει ο κύριος Γιούνκερ ως οι κύριες προτεραιότητές μας που είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης, δημιουργία προσόντων και ικανοτήτων και φυσικά και η κοινωνική προστασία. Πέραν αυτό που είπε ο Βαλδής λοιπόν θα συνεχίσω λέγοντας ότι έχουμε υποσχεθεί να γίνει λειτουργική η πρωτοβουλία για τους νέους. Ένα πράγμα είναι να έχουμε θέσει εργασία, κάτι άλλο είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτε μα και ιδίω οι πιο νέοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι θέσει απασχόληση. Η δική επιτροπή είχε εμπλακεί πλήρω στην διαδικασία προχρηματοδότηση τη πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας για τους νέους. Χαίρομαι και ευχαριστώ τον εισηγητή σας για την ε, πολύ καλή συνεργασία, την ομαλή συνεργασία που υπήρξε μεταξύ των θεσμικών οργάνων χάρη και στην πρότασή σας για να τροποποιηθεί ο κανονισμός του κοινωνικού ταμείου που έγινε πραγματικότητα στις 4 Φεβρουαρίου και τέθη σε ισχύ στις 21 Μαΐου. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, μπορέσαμε πράγματι να εκταμιεύσουμε χρήματα προς τα κράτη-μέρη για την προχρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα προγράμματα για την πρωτοβουλία των νέων. Ένα πρόσθετο ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ είναι στη διάθεση των επιλεξίμων κρατών και περιοχών ώστε πάνω από 600.000 άτομα μπορούν, νέοι μπορούν να υποφελθούν το 2015 και να πρόκειται στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να εφαρμόσουν αυτή την πρωτοβουλία. Έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες μου να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία να παροτρύνουν και να βοηθήσουν προδραστικά τα κράτη-μέλη για να υλοποιήσουν αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά θα σας δώσω μια έκθεση προόδου σε σχέση με την πρωτοβουλία των νέων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχή του 2016 επί τη βάση της πρώτης εκθέσεως αξιολόγησης του προγράμματος για την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι η μακροχρόνια ανεργία. Όπως ξέρετε, η ανεργία μακροχρονίου χαρακτήρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι περίπου 24 εκατομμύρια ατόμων που είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μισή από αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι. Περίπου 30% αυτών είναι άνεργοι για πάνω από δύο χρόνια. Εγώ περατώνω τώρα μια πρόταση για σύσταση σε σχέση με την ενσωμάτωση των μακροχρόνια άνεργων στην οικονομική αγορά. Η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο να αναφέρει και να προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα για αυτή την ομάδα. Με ενδιαφέρει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση της κατάστασης κάθε ανέργου. Τα μέτρα τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν αυτούς τους, την απασχόληση αυτών των ατόμων, τα μέτρα ολοκλήρωσης και υποστήριξη ώστε σε βιώσιμη βάση να μπορέσουν να, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτά θα γίνουν με ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσίας, με μόνο απευθυντικές θηρίδες, όπου οι μακροχρόνια άνεργοι μπορούν να βρουν και απασχόληση. Έχουμε επίση το θέμα της ε, κινητικότητας των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Όπως ξέρετε, η κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικός φορέας αντιμετώπισης της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά συγχρόνως ελοχεύει ο κίνδυνος των καταχρήσεων χρησιμοποιώντας την κινητικότητα αυτή. Γι' αυτό εργάζομαι για ένα πακέτο για την κινητικότητα των εργαζομένων με στόχο να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ενώ παράλληλα εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν τις ε, καταχρηστικές πράξεις από την πλευρά αυτών των εργαζομένων. Το πακέτο αυτό θα περιλαμβάνει και μια πρόταση για ενδεχόμενη ε, αναθεώρηση του κανονισμού για το συντονισμό των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μου αξιολογούν τον αντίκτυπο δυνητικών αλλαγών στους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή και επιπλέον το πακέτο αυτό, η δέσμη μέτρων που θα πρέπει να εγκριθεί στο τέλος του χρόνου θα περιλαμβάνει στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε καλύτερα οποιοδήποτε παραθυράκι το οποίο οδηγεί σε καταχρηστικές πρακτικές ή κοινωνικό dumping. Ένα τέταρτο στοιχείο έχει να κάνει με τα προσόντα και τις δεξιότητες των αυτών που ψάχνουν για εργασία. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δεξιότητες για την ανταγωνιστικότητα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν καταστρεφεί χιλιάδες, εκατομμύρια μάλλον θέσεις εργασίας και πολλοί έχουν αναγκαστεί να δουλέψουν σε εργασίες χαμηλότερων δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση για τα προσόντα και τι δεξιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ορισμένε εξελίξει πρωτοβουλίε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τι δεξιότητε και τα προσόντα τη εργατική μα δύναμη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή <clears throat> Συμμαχία για τι μαθητείε και το πλαίσιο ποιότητο για τι μαθητείε που δίνει μια νέα όθηση στην απόκτηση προσόντων. Θέλουμε επίση να ενισχύσουμε την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουμε τι ευκαιρίες απόκτηση θέσεων εργασία θα υπάρξει μια ειδική σύνοδος των αρμοδίων υπουργών στο άτυπο Συμβούλιο της Ρήγας στις 22 Ιουνίου σε σχέση με συγκεκριμένα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε και θα λάβει χώρα και μια συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου για την επανεκκίνηση της συμμαχίας για τη μαθητεία. Με ρωτήσατε πολλές φορές τι ε, πρέπει να κάνουμε για του, τα άτομα με αναπηρίες. Πρέπει να άρουμε τα εμπόδια ε, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί ε, στην ε, ενιαία αγορά. Είναι κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερος. Ξέρετε ότι υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη γύρανση ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Είναι πρωτογενούς και πρωταρχικής σημασίας για την κοινωνία μας. Αλλά και για την οικονομία μας τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίε να είναι προσβάσιμα από όλους. Για τον λόγο αυτό η, Κομισιόν, η τρέχουσα Κομισιόν εξετάζει να υπάρξει νομοθεσία περί προσβασιμότητας που θα άρει τους φραγμούς μεταξύ κρατών μελών λόγω των διαφορετικών εθνικών κανόνων σε σχέση με την προσβασιμότητα για ορισμένα προϊόντα και για ορισμένε υπηρεσίε. Αυτή η απέτηση λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι σειρές, μάλλον οι ευρωπαϊκές απαιτήσει έχουν σαν αποτέλεσμα να δίνουν στις εταιρείες την δυνατότητα να ξεπερνούν τα εθνικά σύνορά τους και αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο λειτουργική και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά. Αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να καλύψουμε ε, την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών και θα εξασφαλίσουμε την πλήρη και ίση συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες στην ε, οικονομία και στην κοινωνία. Επέκεινα τώρα το 2015, το 2016 θα έχουμε μια σειρά από δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται για του χρόνου. Πρόκειται για την άσκηση refit και την αναθεώρηση των οδηγιών μας σε σχέση με τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, τα προβλήματα ασφάλειας και επαγγελματικών ασθενειών στον χώρο εργασίας και την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Θα φέρουμε κατά πόσα πιθανότητα προτάσει του χρόνου. Σα υπενθυμίζω ότι ο στόχο μα είναι να εξυγχρονίσουμε και να απλοποιήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε θα διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων και προστασία των εργαζομένων, ενώ συγχρόνω διευκολύνουμε την συμμόρφωση και την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στην αναθεώρηση <clears throat> του 2020 Στρατηγική Ευρώπη 2020. Παραμένει αυτό στην ημερήσια διάταξη και θα παρουσιαστεί στο τέλος του χρόνου αυτή η αναθεώρηση. Προς το παρόν οι σκέψεις μας παρακολουθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και έχουν σαν κύριο στόχο να παραμείνουμε πιστοί στους τεθέντες στοχούς σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά επιτεύξιμα που θα πρέπει να είναι οι αιστείες της προσπάθειάς μας και για να στείλουμε επίσης ένα σαφές πολιτικό μήνυμα σε σχέση με τις επιδιωκόμενες προτεραιότητες τα μέσα για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μπορεί να πρέπει να τροποποιηθούν. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα διάλογο ενώπιόν μας και επομένως θα ήθελα να ακούσω τις δικές απόψεις, τις δικές σας ανησυχίες και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα λοιπόν για πολύ σύντομες ε, ερωτήσεις θα ε, ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στους ε, συντονιστές και θα περιμένω τις ε, απαντήσεις αμέσως από εσάς. Ερώτηση-απάντηση, ένα είδος πονκ θα γίνει εδώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Κάστα, ο οποίος είναι συντονιστής του ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε και κυρία Επίτροπε, κυρία Τάισεν. Η πρώτη ερώτησή μου αφορά στον Επίτροπο Ντομπρόφσκι. Ε, πρόκειται για το ε, διαδικασία εξαμήνου του 2015 πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, Έχουμε δει λοιπόν κάποια βελτίωση κυρίως όσον αφορά τους κύκλους των εξαμήνων κατά τα προηγούμενα έτη. Τώρα λοιπόν είναι αυτή η διαδικασία, περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία και έχει στόχο να συμπεριλάβει την ανάπτυξη. Πιστεύω όμως ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα. Όπως είπατε προηγουμένως, παραδείγματος χάρη, τις συστάσεις αναχώρα ε, να γίνουν περισσότερα στον τομέα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Και διερωτώ κατά πόσον ο κύριος Ντορμπρόψκι ενδιαφέρεται να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία στους δείκτες κοινωνικής ε, ε, στους κοινωνικούς δείκτες και στους δείκτες απασχόλησης. Και όσον αφορά την Επίτροπο κυρία Τάισεν, με ενδιαφέρει να μας πει τι ακριβώς ε, συστήνει σε σχέση με τη μακροχρόνια ανεργία. Είπατε προηγουμένως ότι καταθέσατε τις δικές σας ε, συστάσεις, με μεγάλη χαρά λοιπόν. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας, τις προσωπικές συστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κάζα. Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στο ρόλο των ε, κοινωνικών δικτών και των δικτών απασχόλησης και εγώ όσο και η Επίτροπος ε, κυρία Τάισεν επιληφθήκαμε του θέματος αυτού ευθύς εξ αρχής και στόχος μας είναι να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στους δείκτες αυτούς κυρίως οποτεδήποτε αποφασίζουμε για οικονομικές πολιτικές ή οποτεδήποτε αποφασίζουμε για ε, συστάσεις ανά χώρα. Και νομίζω ότι αυτό ήδη αντικατοπτρίζεται στις συστάσεις που έχουμε καταρτήσει. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα από αυτού κατά τον επόμενο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για φέτος, παραδείγματος χάρη, δώσαμε μεγαλύτερη σημασία στις ε, ανασυστάσεις χώρα ε, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει περισσότερο στο να αντιμετωπίσουν οι χώρες τις κοινωνικές ε, προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες, συνεργαζόμαστε και με τον Επίτροπο Μοσκοβισή για να προβάλλουμε περισσότερο τους ε, δείκτες απασχόλησης ε, κάτω από μακροοικονομικό πρίσμα. Όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία, θέλω να σας πω ότι θέλουμε το εξής, όπως ε, και στο, στο μέσο εγγύηση για τους νέους, αυτό που ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους μακροχρόνια άνεργους, γιατί τους ανθρώπους αυτούς δεν τους ενδιαφέρει μόνο να βρουν θέση απασχόλησης, προφανώς και τους ενδιαφέρει και αυτό, αλλά τις περισσότερες φορές τους μακροχρόνια άνεργους, ήδη το 1 τρίτο εξ αυτών δεν έχει εργασία για πάνω από δύο χρόνια. Έχουν λοιπόν προβλήματα στο νοικοκυριό τους, στο σπίτι τους, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Άρα δηλαδή εμείς επιθυμούμε οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι ολοκληρωμένους και να μπορούμε να τους προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων όπου πράγματι θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Και αυτό είναι ένα τμήμα των συστάσεων τις οποίες και επεξεργαζόμαστε. Η κυρία Γιούτα Στάινρουκ, η οποία είναι συντονίστρια των Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δύο ερωτήσεις. Κύριε Τομπρόφσκε, εσείς και ο κύριος Γιούνκα είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμείτε να ενισχύσετε τον κοινωνικό διάλογο. Βλέποντας λοιπόν τη διοργανική συμφωνία και το περίφημο REFIT και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άλλοι, ότι όχι μόνο δεν ενδυναμώνεται, αλλά αποδυναμώνεται ο κοινωνικό διάλογο. Και τι είδου πρωτοβουλίε, όχι συνέδρια, αλλά πώ ακριβώ θέλετε να ενισχύσει το διάλογο ανάμεσα στου κοινωνικού εταίρους και πώ ακριβώ προτίθεστε να συμπεριλάβετε περισσότερο του εργαζόμενου στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις. Κύριε Τάισεν, μιλήσατε για το Label Mobility Package ε, και επίσης και για την επανεξέταση της οδηγίας περί ε, κινητικότητας για την καταπολέμηση του dumping. Είπατε ότι θέλετε να ενισχύσει τα κράτη-μέλη κατά ε, την ενίσχυση αυτών των κοινωνικών εταίρων. Τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να παρεμποδίσουν με κοινωνικά μέτρα το παράτυπο πολλών ε, μορφών απασχόλησης και τώρα η Κομισιόν ε, κατηγορεί τα κράτη-μέλη για παραβίαση κανονισμών. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερους ελέγχους. Πώς ακριβώς λοιπόν προτίθεται να προχωρήσει η Κομισιόν στο μέλλον. Ο κύριος Ντομπρόφσκι. Ευχαριστώ, ο κύριος Ντομπρόφσκης. για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου για να υπενθυμίσω ορισμένες πρακτικές πρωτοβουλίες που είναι ήδη εν εξελίξη. Ανέφερα την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό έχει γίνει ήδη εφέτος, αλλά έχουμε δώσει περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους στα κράτη-μέλη το ετοιμάσουμε τις ειδικές αναχώρα συστάσεις. Θα συνεχιστεί αυτό επίσης. Ο στόχος μας είναι να εμπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι περισσότερο και σε εθνικό επίπεδο στις συζητήσεις για τις προτεραιότητες ετησίας ανάπτυξης, τις έκθεσης ετησίας ανάπτυξης και την επόμενη φορά θα ζητήσουμε και την ανάδραση των κρατών μελών για το πώς εμπλέκουν τους κοινωνικούς εταίρους σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για την πρωτοβουλία REFIT για, τον, την καλύτερη ρύθμιση την καλύτερη νομοθεσία. Είχαμε μια συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε τη δική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και θα τροποποιήσουμε και τις ε, διαδικασίες μας αιτήσει των κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις αντικτύπου, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις, ώστε να λάβουμε υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο που επέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και για το πώς θα ενισχύσουμε το διμερή διάλογο. Φυσικά ο διμερής διάλογος είναι πρώτα απ' όλα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Μπορούμε να τον διευκολύνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε είναι να εξασφαλίσουμε τον τριμερή διάλογο και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε αυτού του είδους τον διάλογο. Τάισεν, ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω Ολλανδιστή. Ναι. Αν θέλετε πάλι τα ακουστικά, τα ακουστικά σας μου με ρωτάτε τι κάνουμε σε σχέση με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό dumping και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους κατά του dumping αυτού. Πρέπει να διευκολύνουμε από την άλλη πλευρά την κινητικότητα των εργαζομένων γιατί η ενιαία αγορά θα πρέπει να λειτουργεί και για τους εργαζομένους. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αποσπάσεις των εργαζομένων θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καταχρηστικές πρακτικές Είπατε ότι τα κράτη-μέλη παίρνουν κάποια μέτρα. Εμείς έχουμε απευθύνει οχλήσεις σε χώρες όπως είναι πραγματικά η Γερμανία για το, τις ε, ελάχιστες αποδοχές στον τομέα των μεταφορών. Η Γερμανία έχει εισαγάγει ελάχιστο μισθό για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό γιατί αυτό επιτρέπει να αντιμετωπιστεί μια κλιμάκωση προς τα κάτω των αποδοχών Πρέπει λοιπόν να γίνει σεβαστό αυτό, το να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο αποδοχών στον τομέα των μεταφορών. Αυτό το εξετάζει η Κομισιόν, είναι εφικτό πιστεύω για τις διαμεθοριακές ε, υπηρεσίες όταν μιλάμε για καμποτάζ, αλλά όχι όταν μιλάμε για διέλευση, όταν πρόκειται για διεθνείς μεταφορές εν διελεύση. Θα πρέπει εφαρμόζοντας αυτήν την ε, ρύθμιση να έχουμε υπόψη μας και την αρχή της αναλογικότητας. Υπενθύμησαμε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αυτή την αρχή. Περιμένουμε την ε, απάντηση. Αλλά δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη Γερμανία να υιοθετήσει μέτρα αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην εσωτερική αγορά τα μέτρα που αναλαμβάνει κάθε χώρα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα λάβουμε υπόψη μα στο πακέτο για την κινητικότητα εργαζομένων. Εντάξει. Θα σας ρωτήσουν και άλλα. Κύριε Τέρνες, από την ομάδα των φιλελευθέρων. Α, Η κυρία Μακιντάερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και τον κύριο Ντομπρόφσκη και την Επίτροπο Τάισεν θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους, την οποία χαιρετίζω ιδιαίτερα. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε για, τον, για την καλύτερη νομοθεσία. Για μένα η καλύτερη νομοθεσία δεν είναι μια αφηρημένη και ιδεολογική ιδέα είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και είναι η ανάπτυξη η οποία δημιουργεί θέσει απασχόληση. Είναι θεμελιώδες λοιπόν κάτι τέτοιο για το έργο της Επιτροπής Απασχόλησης. Κύριε Ντομπρόφσκης, μιλήσατε για το ανοιχτό πνεύμα και την διαφάνεια στις διαβουλεύσεις. Πρέπει όμως να εστιάσουμε περαιτέρω στις εκθέσεις αντικτύπου εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, σε όλη λοιπόν τη διάρκεια και να δούμε τι επιτυγχάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις συγκεκριμένες ιδέες που έχετε και οι δυο σας για το πώς θα δώσετε συνέχεια στις ιδέες του Προέδρου Τίμερμανς για την καλύτερη νομοθεσία και επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αποκομίσουμε κάποιο αποτέλεσμα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Ελπίζω ότι είσαστε ευθυγραμμισμένοι όλοι οι αντιπρόεδροι, γιατί η κυρία Τζότζεβα είπε ότι πρέπει να υπάρξει σωστή αξιολόγηση τη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Τι επιτυγχάνουμε λοιπόν με αυτή τη χρηματοδότηση. Η Ευρώπη δεν έχει ένα απίθμενο βαρέλι χρημάτων στη διάθεσή τη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά αποδίδουν του καρπού που θέλουμε. Η άλλη πλευρά τη καλύτερη νομοθεσία, και τα είπε και σήμερα το πρωί ακόμα ο κ. Τίμερμαντ στην διακομματική ομάδα για τι μικρομεσαίε, επιχειρήσεις πρέπει να δούμε και τα μη νομοθετικού χαρακτήρα μέτρα. Η απάντηση σε όλα τα προβλήματα δεν είναι μοναχά η νομοθεσία. Θα πρέπει να είμαστε ευφιέστεροι για τον τρόπο αντιμετώπιση των προγραμμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο τι κάνετε για να εξετάσετε μέτρα τα οποία έχουν μη νομοθετικό χαρακτήρα για να επιτύχετε τους στόχους σας. Σε σχέση με την καλύτερη νομοθεσία, όπως είπα και προηγουμένως, η βασική ιδέα είναι όταν γίνεται αξιολόγηση για νέα ε, νομοθεσία, προτού λάβουμε τις αποφάσεις, να προβαίνουμε σε αξιολόγηση αντικτύπου για να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της νομοθεσίας και να γίνεται και δημόσια διαβούλευση, να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και να λάβουμε να ακούσουμε και τις δικές τους απόψεις για την προτινόμενη νομοθεσία. Βάσει λοιπόν της δικής μας κατανόησης, αυτό θα μας επιτρέψει τελικά να έχουμε μία ε, καλύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ε, πιο ενημερωμένη. Πολλές φορές υπάρχουν ε, λανθασμένες αντιλήψεις ε, για την επιπλέον νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην προσπάθεια αξιολόγησης πριν από την νομοθεσία, ώστε όταν προτείνεται μία νομοθεσία, η απόφασή μας να είναι ε, σωστή και εξισορροπημένη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάισεν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά αυτήν ε, την πρωτοβουλία για την καλύτερη νομοθεσία, είναι γεγονός ότι δεν χρειάζεται συνέχεια να νομοθετούμε περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της ότι θα κάνει οικονομία νομοθεσίας, ότι θα επικεντρώνεται περισσότερο στα πιο σημαντικά και στα ζητήματα που επιζητούν μία απάντηση ευρωπαϊκή. Είναι κάτι για το οποίο συμφωνούν όλοι οι Επίτροποι. Δεν υπάρχει στο σώμα των Επιτρόπων ούτε μία αντίρρηση ως προς αυτό. Όσον αφορά τώρα τις μη νομοθετικές ε, δυνατότητες και θα αναφερθώ τώρα στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις εταιρικές ε, σχέσεις επιχειρήσεις και ο χώρος της επικοινωνίας, ε, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ εύκολο, ειδικότερα για τους νέους. Όχι μόνο δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, αλλά εξασφαλίζει ότι οι νέοι έχουν τις σωστές δεξιότητες προκειμένου να εργαστούν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή την πρώτη επαγγελματική εμπειρία που χρειάζονται οι νέοι δεν μπορούν να την έχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μαθητεία και άσκηση. Για μένα οι εγγυήσει των νέων για τους νέους πρέπει να προωθηθούν, πρέπει να τις ενισχύσουμε. Πρέπει να πάμε όμως και επιτόπου εκεί όπου υπάρχουν τα προβλήματα να δημιουργήσουμε μια δυναμική για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου όχι υποχρεωτικά νέους νόμους, όχι υποχρεωτικά ε, νέους κανόνες, αλλά να δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ ατόμων ε, με καλή ε, θέληση που θέλουν να επιφέρουν αποτελέσματα. Κυρία Μάκιντάιρ, μερικοί πιστεύουν ότι η δράση μπορεί να περάσει μόνο από νέα νομοθεσία, όμως μπορεί να γίνουν πράγματα επιτόπου που ε, τα περιμένουν οι πολίτες, γιατί αυτό που περιμένουν οι πολίτες είναι αποτελέσματα και αυτό θέλουμε να κάνουμε και ε, βάσει αυτών θέλουμε να κρυφθούμε σε πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ τρία ερωτήματα πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο έχει να κάνει με την οδηγία για τη μετρική άδεια ή τη γονική άδεια. Ξέρουμε ότι αυτό είναι μια αρμοδιότητα ε, που αντιμετωπίζεται από άλλους συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τη μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας και θα ήθελα να ξέρω αν θα υπάρξει μια νέα πρόταση της Κομισιόν, αν έχετε κάποιες ε, προθέσεις σε σχέση με το σημείο κίνησης αυτής της πρότασης σε συγκεκριμένο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα επίπεδα προστασίας των γυναικών, των μητέρων. Δεύτερον, για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεότητα. Το ερώτημα είναι το εξή. Είναι φυσικά θετικό το ότι μπόρεσε να υπάρξει μια προχρηματοδότηση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόγραμμα. Αναρωτιέμαι όμως αν υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες να αυξήσουμε τα προτινόμενα, τα προβλεπόμενα ποσά για αυτό το πρόγραμμα. Και τρίτον, έχει να κάνει το τρίτο ερώτημά μου με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την μαθητεία επαγγελματικού χαρακτήρα που ουσιαστικά είναι επιδοτούμενες φτηνές θέσεις εργασίας που καλύπτουν άλλες θέσεις εργασίας που έχουν καταστραφεί από την κρίση. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και για τους άνεργους που χάνεται η θέση εργασία τους, αλλά και για τους νέους οι οποίοι περνάνε από τη μία μαθητεία στην άλλη χωρίς να έχουν καμία απολύτως πρόπτικη για το μέλλον. Πώς θα παρακολουθήσετε και θα εποπτεύσετε μέσα στο πρόγραμμα εγγύησης για το νέο τέτοιου είδους καταστάσεις και πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν οδηγούν σε ατέρμονες μαθητείες και ότι θα οδηγήσουν όλα αυτά σε μόνιμες θέσεις εργασίας και δεν θα κατασταθούν αυτές τις θέσεις εργασίας για πάντα. Κύριος Μουλαύσκης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας. Καταρχήν όσον αφορά την πρώτη ερώτηση θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί υπήρξαν ουσιαστικές προσπάθειες κυρίως κατά τους τελευταίους μήνες να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όσον αφορά την άδεια μητρότητας. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε επ' αυτού και η δική μας η δέσμευση είναι ε, να προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση. Αν τελικά δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία, θα αποσύρουμε αυτή την πρόταση και θα καταθέσουμε μια νέα καινούρια ε, που ε, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί. Όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους, τώρα εστιάζουμε την προσοχή μας την ε, ε, εφαρμογή της υπάρχουσας εγγύησης και με βαρύ μορφή, όπως ανέφερε και η Επίτροπος, δηλαδή μεταφέρεται στα κράτη-μέλη. Εμείς, το έχω πει αρκετές φορές, ε, είμαστε ανοιχτοί στο να επεκταθεί αυτή η πρωτοβουλία, να συμπεριλαμβάνει και άλλες μορφές ε, χρηματοδότησης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή ε, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να καταστεί λειτουργική αυτή η εγγύηση. Η συνάδελφός μου, κυρία Τάισεν, έχει το λόγο. Όσον αφορά την πρωτοβουλία για τους νέους θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα και θέλω να πω στους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο ότι και το κοινωνικό ε, ταμείο έχει χρήματα, τα οποία, η κονδύλια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη μορφή ε, πρωτοβουλίας. Υπάρχουν ε, τα στοιχεία από το ελεγκτικό συνέδριο, 1,5 δις για 7 χρόνια. Αυτά μπορούν να εκταμιευτούν για λειτουργικά προγράμματα έτσι ώστε οι νέοι να αποκτήσουν θέση απασχόλησης. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία όταν θα ολοκληρωθεί και δεν είναι ότι θα σταματήσει κάποια στιγμή ξαφνικά. Υπάρχουν μακροχρόνιες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Εν πάση περιπτώσει, ήδη κατά το 2015 θα εξετάσουμε και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα κονδύλια. Όσον αφορά τα στάζ, τις μαθητίες, ε, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα ε, και γνωρίζουμε ότι οι νέοι οποτεδήποτε βρίσκουν θέσεις απασχόλησης, αυτές απασχόληση. Αυτέ είναι επισφαλίσει ένα είδος ε, στάζ ή ή ένα μαθητείας, είναι συμβάσεις έργου, μορφέ απασχόλησει με σύμβαση έργου. Η ενα ειδο μαθητειας ειναι συμβασει εργου μορφε απασχολησης με συμβαση επιμένει και στι ε, συστάσεις ανά χώρα να βρεθεί κάποια άλλη δυνατότητα απασχόλησης και βλέπετε, αν δείτε αυτές τις συστάσεις θα δείτε ότι εμείς επισημαίνουμε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Ε, υπάρχουν πολίτες και εργαζόμενοι που προστατεύονται θαυμάσια, αλλά για άλλους δεν υπάρχει καν η δυνατότητα να ενταχθούν ε, στην αγορά εργασία και αν τότε αποκτούν μόνο συμβάσεις έργου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε ότι αυτό ίσως είναι μια καλή λύση, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και αυτό στο διηνεκές. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την ε, κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Κατά τα άλλα, όταν γίνεται λόγος για στάζ και για μαθητείες, είναι σαφές ότι εδώ πρέπει να υπάρχει καλή ποιότητα. Το θέμα δεν είναι να παρκάρει και κανείς τους νέους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά να υπάρχει κοινωνική προστασία και να τους προσφέρεται η δυνατότητα να βελτιώσουν και τις δεξιότητές τους κατά διάρκεια αυτής της μορφής εκμάθησης για να μπορούν να ανταχθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Λάμπερτ ε, που είναι συντο... στην κυρία Λάμπερτ που είναι συντονίστρια. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στρατηγικής ε, σημασίας αφορά όλο αυτό το θέμα των πράσινων θέσεων απασχόλησης, το θεματολόγιο για χαμηλές εκπομπές ε, καυσαρίων του άνθρακα, για την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει κάποιες ε, δεσμεύσεις σχετικά με την μετάβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης. Ε, σε αυτό το πλαίσιο θα τοποθετηθώ. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα της απασχόλησης τι ακριβώς προτείνει, τι θα προτείνει σε αυτές τις συζητήσεις στο Παρίσι αλλά και γενικότερα εδώ στις, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς θα ενταχθεί όλο αυτό και στη στρατηγική για τις δεξιότητες. Δηλαδή, θα αναζητήσουμε δεξιότητες που να ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή θα μιλάμε έτσι γενικά για δεξιότητες όπως γίνεται στις συστάσεις αναχώρα, στο περιφερειακό προγραμματισμό και το καθεξής. Και όσον αφορά τους κοινωνικούς εταίρους γνωρίζουμε ότι η ουσιαστική συμμετοχή τους μέσα στις εταιρείες έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές ε, στην αποτελεσματικότητα των πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό πώς ακριβώς εντάσσεται στον κοινωνικό διάλογο. Ο κύριος Ντομπρόφσκι. Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από το 2013 και αυτή υπογραμμίζει το ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πράσινες θέσεις απασχόλησης αλλά και να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί και το πράσινο θεματολόγιο. Αυτό το ε, στοιχείο πρέπει να συμπεριληφθεί περισσότερο στο, στο δική μας τη δέσμη μέτρων. Όσον αφορά τώρα ε, συστάσεις αναχώρα, ε, να σας πω τι κάναμε. Εμείς επιλέξαμε να υπάρχουν λιγότερες αλλά πιο στοχευμένες τέτοιου είδους συστάσεις οι οποίες εστιάζονται στα κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Άρα δηλαδή δεν θα έχουμε εφέτος συστάσεις αναχώρα για θέματα ενέργειας. Δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις με θέματα τα οποία καλύπτονται από άλλους τομείς. Ας πούμε τα θέματα της ενέργειας μπορούν να ε, αντιμετωπιστούν με έγγραφα που αφορούν στην Ενεργειακή Ένωση. Τώρα για τους στόχους ε, του 2020 Πράγματι, αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν στο θεματολόγιό μας. Εργαζόμεθα για να τους επιτύχουμε και επίσης επεξεργαζόμεθα και μία αναθεώρηση της στρατηγικής του 2020 σχετικά με τις εκπομπές διοξυδίου του άνθρακα. Εκεί η στόχοι είναι κάπως καλύτερη σε σχέση με άλλους που αφορούν ε, στην απασχόληση, παραδείγματος χάρη. Η κυρία Τάισεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων απασχόληση, αυτή μεταβάλλεται. Οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει κανείς εργασία, το έχω ήδη πει, έχουν αλλάξει. Πάρα πολλές ε, θέσεις έχουν καταργηθεί λόγω κρίσης και θα εμφανιστούν νέες. Και αυτό έχει σχέση και με τη διαφοροποίηση οικονομίας. Και η οικονομία θα αλλάξει και έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Άρα δηλαδή οι δεξιότητες είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, ένα θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να λειτουργεί η οικονομία και οι νέες θέσεις απασχόλησης ε, ε, να βρουν και αυτές ένα χώρο μέσα στην οικονομία. Αυτό έχει μπει ε, στο θεματολόγιο για τις δεξιότητες. Το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλουμε να το προάγουμε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά πετούν την προσοχή μας όπως επίσης και το ότι αλλάζουν εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τώρα στις ε, δεξιότητες, δεν μπορούμε να πούμε επακριβώς τι θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη και από τις ε, περιφέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν λέμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην επαγγελματική ζωή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι απαραίτητο έτσι ώστε να διευκρινιστεί ποιε είναι οι απαραίτητες δεξιότητες. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Πάρα πολύ θα ήθελα να σας λόγο στη Λάρο Άγκια που είναι συντονίστρια του FDD, του κόμματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και την κυρία και τον Επίτροπο και την κυρία Τίσεν. Για τον κύριο Ντομπρόφσκι, να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, θέλω να σα ρωτήσω, μήπως μπορείτε να σχολιάσετε ποιε είναι οι οικονομικές προβλέψεις της άνοιξη, κυρίως όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στα σωρευμένα στοιχεία για την απασχόληση στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης σε αυτά και στα άλλα που είναι εκτός Ευρωζώνης. Μήπως μπορείτε να μας τα σχολιάσετε αυτά τα στοιχεία. Σήμερα το πρωί ο συνάδελφος ε, Τίμερμανς μίλησε για το Refit, για καλύτερη νομοθεσία, ε, οξυγόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για την ανάπτυξη. Ωραία λόγια, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις που να αφορούν το Refit και αν ναι, ποιες είναι οι ενδείκτες. Συγκεκριμένα ερωτώ, τι προτίθεστε να κάνετε. Πάω τώρα στον κοινωνικό διάλογο. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι συμφωνεί ότι θα υπάρξει βοήθεια στην Ελλάδα και αμέσως προκύπτουν διαψεύσεις. Εμείς πολίτες είμαστε και θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει γιατί μιλήσατε για την εγγύηση για τους νέους. Στην Ιταλία, ξέρετε, απέτυχαν όλα αυτά και μάλιστα πρόκειται και δυσαρέσκεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να σας πω κάτι, δεν το λέω εγώ, το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Σήμερα το πρωί ε, θα συναντηθούμε με το ελεγκτικό συνέδριο, η οποία μας κατηγορεί και λέει ότι είμαστε ένας από τους χειρότερους χρήστες αυτών των εργαλείων. Ούτε τα απασχόλησης ε, δημιουργήσαμε, ούτε αποτελεσματικά εργαλεία. Και μάλιστα σήμερα ε, στον Ιταλικό τύπο διαβάζει κανείς ότι ο ΣΑ μας επιπλήττει για πολλωστή φορά και γιατί λέει ότι οι Ιταλοί νέοι ε, είναι άνεργοι αλλά δεν έχουν και δεξιότητες και αυτοί που δεν έχουν δεξιότητες δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Αυτό το λέει ε, ο ΣΑ και όχι το κίνημα των πέντε αστέρων, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους, κατά την άποψή μου, το θέμα είναι από πού ξεκινάμε και πού φτάνουμε. Κύριε Επίτροπε, ο κύριος Επίτροπος ε, είπατε ότι θα ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη να μας πούνε για το πώς μπορούν να διαβολευτούν με τα κράτη-μέλη και σας παρακαλώ πολύ να επιλέξετε ε, τα κράτη-μέλη εκείνα που είπαν ότι θέλουν να διαβολευτούν γιατί αν δείτε ας πούμε το πώς έγινε η σχολική μεταρρύθμιση στην Ιταλία με την ε, ε, συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Ε, εκεί τι να σας πω, ούτε καν υπήρξε αποτελεσματική διαβούλευση και οι κοινωνικοί εταίροι, να σας το πω απλά, θεωρούν με απλά λόγια ότι τους δουλεύουν. Αν θέλετε, τους εξαπατούν. Ο κύριος, ο κύριος <clears throat> βεβαίως λέει ο κύριος Βαλδής. Πολλές ερωτήσεις θα σας απαντήσω σε ένα λεπτό βέβαια. Πρώτα απ' όλα, για τα, τις οικονομικές προβλέψεις. Είναι ιδιαίτερα σαφές ότι οι αρινές οικονομικές προβλέψεις βλέπουν βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης 1,8 για την περιοχή του ευρώ. 1,5 για την περιοχή του ευρώ και 1,8 για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε επίσης μείωση της ανεργίας και στην περιοχή του ευρώ και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτά τα οποία <clears throat> βλέπουμε είναι μείωση στα 11,3 στην περιοχή του ευρώ και 9,8 στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με πέρσι είναι σαφής η φθήνουσα τάση και στην περιοχή του ευρώ αλλά και στην Ευρώπη των 28. Φυσικά ποικίλει μεταξύ κρατών μελών αυτή η εικόνα. Είναι σημαντικά διαφορετικές οι, τα επίπεδα ανεργίας, αλλά δεν λέω ότι υπάρχει απόκληση μεταξύ της περιοχής του Ευρώπη και της υπόλοιπης Ευρώπης και στις δύο περιοχές μειώνεται η ανεργία. Για την πρωτοβουλία ρίφη και πάλι. Εδώ πρόκειται περισσότερο για την διαδικασία λήψης αποφάσεων με την ιδέα ότι οι ιδέες προτού οδηγηθούν σε αποφάσεις θα πρέπει να περνάνε από μια διαδικασία ελέγχου αντικτύπου και διαβούλευσης προτού προχωρήσουν προς την επίσημη λήψη αποφάσεων. Πρωτού οι πρωτοβουλίες αυτές φτάσουν στο τελικό σημείο τους. Να υπάρχει λοιπόν περισσότερη διαβούλευση πριν ληφθούν αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριε Τάισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι στη χώρα σας η ανεργία μακροχρόνιου χαρακτήρα είναι πολύ υψηλή. Αν δούμε το επίπεδο κατάρτισης του πληθυσμού στην Ιταλία, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία έχουν άτομα τα οποία έχουν δίπλωμα βάθμιση εκπαίδευσης. Δεν μπορεί η πρωτοβουλία για τους νέους να λύσει όλα τα προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη. πρέπει να γίνουν διαφορετικέ αλλαγέ για να δημιουργηθούν δομές οι οποίε είναι πιο ευεπίφορε για την ολοκλήρωση τη αγορά εργασία και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά εργασία, Εδώ με την πρωτοβουλία για την νεότητα μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους και να έχουμε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα αυτό. Για την Ιταλία λοιπόν παρακολουθούμε την κατάσταση όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μονάχα θέμα παροχής ε, κονδυλίων αλλά και παρακολούθησης για να εξασφαλίσουμε ότι οι δικαιούχοι έχουν υποστηριχθεί, να δούμε τι έχει επιτευχθεί, τι αλλαγές έχουμε επιτύχει στο χώρο εργασία με τη χρηματοδότηση αυτή. Αν κάποιο έχει υποφεληθεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μετά από 6 μήνες αυτό έχει οδηγήσει σε μια θέση εργασία ή όχι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση θα πρέπει να το ξέρουμε. δεν βγάζουμε από το καπέλο τα στοιχεία. Έχουμε ενδείκτες οι οποίοι έχουν εγκριθεί από μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνουμε υπόψη και ποιοτικά στοιχεία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η εγγύηση για τους νέους θα χρησιμοποιηθεί σωστά, θα κατευθυνθεί με τον καλύτερο τρόπο ενδεχομένως να αλλάξει η στόχευσή της αν χρειάζεται, χάρη και στις ειδικέ αναχώρα συστάσεις. Μην περιμένετε θαύματα μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο. Αλλά μπορείτε να περιμένετε πρόοδο, όλα μπορούν να επιτευχθούν. <clears throat> χρειάζεται όμως πρόοδος, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες στους νέους για να βρουν τη θέση απασχόλησης. Υπάρχουν πολλά ονόματα τώρα από τους υπόλοιπου ομιλητές. Έχουμε τις ψηφοφορίες που πρέπει να γίνουν μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων. παρακαλώ να είσαστε σύντομοι ερωτήσεις ενός λεπτού και αποφασίστε ρωτά τον κύριο Ντομπρόφσκης ή την κυρία Τάισεν. Θα έχετε μετά πολύ σύντομες απαντήσεις και θα προσπαθήσουμε να, διεξα... να διεξέλθουμε όλο τον κατάλογο. Δεν σας το υπόσχομαι θα γίνει αυτό. Μωράν Σατιέ, Ιαγγέλιους, Μαν, Ριφάι, Μπέκερ. Eh, Balas, eh, Sander, Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Sojdorova, and Pirinsky. Anybody missing? Okay. That means that... Αυτό σημαίνει, ναι. Παρακαλώ, ένα, σε ένα επίτροπο θα απευθυνθείτε και θα μιλήσετε για ένα λεπτό. Η κυρία Μόρια Σαρτιέ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας πω Ευχαριστώ καταρχάς. Ευχαριστώ για την αποτελεσματικότητα, για την προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για τους νέους. Εάν η Ευρώπη ανακτήσει την εμπιστοσύνη της, θα το κάνει με την αποτελεσματικότητα ε, μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων. Τρεις μήνες μας είπατε ε, μας είπατε για τα κονδύλια ότι ε, ε, στα κράτη-μέλη την Παρασκευή. Πρέπει να εμπνευστούμε από αυτή την αποτελεσματικότητα ε, για να εμπνεύσουμε και εμπιστοσύνη στους πολίτες στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου αφορά τους νέους ε, ηλικίες μεταξύ 25 και 30. Ξέρετε ότι όταν ε, ιδρύσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαμε παρατηρήσει ότι υπήρχαν τόσοι άνεργοι μεταξύ 25 και και 30 ε, και, και μεταξύ 15 και 25. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για αυτή την ομάδα πληθυσμού. Μιλάμε συνήθως για νέους ε, που ε, μένουν στο πανεπιστήμιο, καθυστερούν τις σπουδές τους, αλλά μετά δεν βρίσκουν θέση εργασίας. Δεύτερο ερώτημα, για αυτό που είπατε για τις ικανότητες και τις δεξιότητες. Πώς μπορούμε αυτές, αυτά να ε, τα χρησιμοποιήσουμε, τα αξιοποιήσουμε σε σχέση με την εμπειρία των νέων. Πρέπει να αλλάξουμε και την οτροπία στον τομέα της ε, Εκπαίδευση αλλά και στο Europass. Τρίτον, ε, η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, πώς μπορούμε την έρευνα και την ανάπτυξη να την αξιοποιήσουμε προς όφελος της ένταξης ε, των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λεπτά. Μην το ξανακάνετε. Μην το κάνετε οι υπόλοιποι. Η κυρία Τάισεν. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, σύντομη. Με δύο λόγια, κυρία Μωράν Σαφία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για την προχρηματοδότηση και να βελτιώσουμε την προχρηματοδότηση για τις εγγύησεις για την νεολαία. <coughs> Πρέπει να κάνουμε μια συλλογική δουλειά μαζί με το Κοινοβούλιο και μόνο χάρη σε αυτή τη συλλογική δουλειά μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Οπότε συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ πολύ. Δεξιότητε, ικανότητε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι γεγονό ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στου νέου για να έχουν μια πρώτη εμπειρία. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα. Οι επιχειρήσει πρέπει να καταλάβουν ότι οι νέοι δεν βγαίνουν από την εκπαίδευση έτοιμοι να δουλέψουν τουλάχιστον στην επαγγελματική ε, κατάρτιση πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Δεν οδηγεί αμέσως σε θέση εργασίας. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις επαφές μας με τις επιχειρήσεις, να υπάρξει συνεργασία, ώστε οι άνθρωποι που βγαίνουν από την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση να είναι πιο πολύ πιο έτοιμοι να δουλέψουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν μαθητείες επιχειρήσεις, ε, άσκηση, ε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γενικευθούν. Έρευνα Καινοτομία, ναι, συμφωνούμε απολύτως και έχουμε υπόψη μας αυτήν ε, την νομοθεσία για την προσβασιμότητα, για τη βελτίωση των επιχειρήσεων και να υπάρχει επίση επίσης εναρμόνιση. Πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των ε, ε, διαφόρων φορέων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, περισσότερος ανταγωνισμός, περισσότερη έρευνα, περισσότερα προϊόντα καλύτερης ποιότητας και πιστεύουμε ότι χρειάζεται εξέλιξη για άτομα που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα, προβλήματα ας πούμε προσβασιμότητας. Και με το σχετικό νόμο ελπίζω ότι θα δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιονκέριους. Θα θέσω το ερώτημά μου στα Ολλανδικά για να μιλήσω πιο γρήγορα. Προς την Επίτροπο Τάισεν το ερώτημά μου. Υπάρχουν προτάσεις στο πλαίσιο ε, του REFIT υπήρχε διοργανική συμφωνία. για τη μείωση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να λαμβάνουν αποφάσεις, εσείς θα αντιταχθείτε σε αυτό. Επίσης άκουσα ότι υπάρχουν και προτάσεις ε, γύρω από το πακέτο της κινητικότητας των εργαζομένων με προτάσεις για το συντονισμό των πολιτικών ε, ε, κοινωνικού χαρακτήρα. Εγώ είμαι αρκετά απογοητευμένη από αυτά που έχουν εξαγγελθεί, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, πρέπει να γίνει πιο εντατική η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να μην υπάρχουν παραθυράκια νομοθετικά και γι' αυτό πρέπει να νομοθετήσουμε. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι τέτοιο. Και τελευταίο ερώτημά μου. Γνωρίζετε ότι έχουμε μία ακρόαση κατόπιν έκθεση του Πανεπιστημίου της Γάνδης για τον τομέα της αεροπορίας υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές πρακτικές κοινωνικού και Έχετε σκοπό να κάνετε συγκεκριμένα για αυτό τον τομέα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιονγκέριους, για το πρώτο που είπατε, ξέρετε ότι ο κύριος Ντομπρόφσκης μαζί με τον κύριο Τίμερμανς και εγώ Ήρθαμε σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους, μιλήσαμε και στην άτυπη σύνοδο της, ε, στη για το κοινωνικό ντάμπινγκ και έχουμε και, αυτό, και αυτή την πρωτοβουλία της καλύτερης νομοθεσίας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα επιτύχουμε όλα αυτά, το είπατε κι εσείς. Υπάρχουν συμφωνίες που πέρασαν ε, αυτόνομα από τους κοινωνικούς εταίρους. Τι πρέπει να κάνουμε πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάναμε για την νομοθεσία, που κάναμε για τη διαβούλευση και στην νομοθεσία, γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, υπάρχουν θέματα τα οποία ε, αφορούν συγκεκριμένα τους κοινωνικούς εταίρους και νομίζω ότι συμφωνούμε όταν λέμε ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, ότι πρέπει ε, ο, ο κοινωνικός χαρακτήρας των προβλημάτων να, ε, το, του διαλόγου να ενισχυθεί μέσω δημοσίων διαβουλεύσεων όσον αφορά αυτών των ε, ε, αποφάσεων που λαμβάνουν ε, μονομερώς οι κοινωνικοί εταίροι. Όσον αφορά τώρα το πακέτο για την απόσπαση των εργαζομένων και την κινητικότητα. Κοιτάξτε, δεν έχει ληφθεί απόφαση, δεν υπάρχει τίποτε το τελεσμένο, ούτε για αυτό που θα κάνουμε, ούτε για αυτό που δεν θα κάνουμε. Δεν έχουμε Έχουμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά το συντονισμό των κανόνων ε, ε, τώρα. Το τι θα κάνουμε στο πλαίσιο συγκεκριμένα αυτής της οδηγίας για την απόσπαση δεν το ξέρω. Σας το λέω ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν έχουμε αποφασίσει ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αν το Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο βελτίωσης της ε, τρέχουσας νομοθεσίας, ευχαρίστω να έρθετε σε επαφή μαζί μας γιατί ε, και εμείς ακόμη το συζητούμε όσον αφορά τώρα την αεροπορία που θέσατε συγκεκριμένο ερώτημα, γνωρίζω τα προβλήματα ε, οι υπηρεσίες μας έχουν πραγματικά αρχίσει να ασχολούνται πολύ εντατικά με αυτό το θέμα και το συζητάμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα σχετικά προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Κοιτάξτε, μιλήσαμε μόνο, μόλις για την παραβίαση των συνθήκων, κυρίως στην οδηγία περί απόσπασης εργοζομένων. Ε, το θέμα έχει εξεταστεί στις ε, αεροπορικές εταιρείες, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις όπου αναφέρθηκε ότι δεν είστε αρκετά κινητικοί, πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή και φτάνουμε και μέχρι την επιστολή του ε, τεχνίτη και μέχρι του να μπορούμε όμως να διεξάγουμε ελέγχους. Τι θέλουμε τελικά να κάνουμε, θέλουμε να αποκαλύπτονται οι παράτοπα εργαζόμενοι, θέλουμε σε περίπτωση που υπάρχει ατύχημα οι άνθρωποι να προστατεύονται. Και ε, το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να υπονομεύσουμε την εσωτερική αγορά. Αυτή η πίεση για την απόλυτη κινητικότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει βασικά να διατηρήσουμε την ποιότητα που αμφισβητείται. Όλοι θέλουμε την κοινή αγορά και κοινού κανόνες, αλλά δεν επιθυμούμε αυτό το οποίο επιτύχαμε στο επίπεδο της ποιότητας να αμφισβητείται από τους κοινωνικούς εταίρους. Και νομίζω ότι η Επίτροπος μας που είναι αρμόδια για κοινωνικά θέματα δεν έχει δηλώσει προσιλωμένη σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ κύριε Μαν. Αγαπητέ Θωμά, συμμερίζομαι τι ε, <clears throat> ανησυχίε σα και νομίζω ότι συμφωνούμε για το επίπεδο φιλοδοξία που πρέπει να τρέχουμε για την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να λειτουργήσει. Έχουμε αξίε στην Ευρώπη, κοινωνικέ αξίε. Θέλουμε την οικονομική πρόοδο, αλλά θέλουμε και την κοινωνική πρόοδο που είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και τα δύο στοιχεία λοιπόν το κοινωνικό και το οικονομικό είναι αλληλένδετα. Αυτό είναι ο άξονα που ακολουθεί η Κομισιόν. Τώρα, όταν λαμβάνουμε αποφάσει, εμεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι αποφάσει αυτέ <clears throat> να συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ελάχιστο μισθό στη Γερμανία είναι ένα θετικό στοιχείο και φυσικά μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα στον τομέα των μεταφορών, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ε, καταγγελίες που έχουν γίνει και να δούμε αν σε νομικό επίπεδο μπορεί να ευδοκιμήσει αυτό το μέτρο. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στο φως των Ευρωπαϊκών Συνδικών και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία διαβιβάστηκαν και στις γερμανικές αρχές. Δύο μήνες έχουν για να απαντήσουν ενδιάμεσα, στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα. Έχουν ανασταλεί τα μέτρα αυτά στον τομέα των μεταφορών. Συνεχίζει το διάλογος. Θέλουμε η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει και τα κράτη-μέλη έχουν φυσικά και τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπενεφάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε Τάισεν, λόγω της οικονομικής κρίσης ο αριθμό των παιδιών που βρισκόνται σε κίνδυνο ένδυαση ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 εκατομμύριο βάσει τη Eurostat 26,5 εκατομμύρια παιδιά στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύουν να πέσουν σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού ή ενδίας. Εμεί ω σοσιαλιστέ είμαστε προσιλωμένοι στον αγώνα κατά τη παιδική ένδυα και θέλουμε να έχουμε μια εγγύηση για τα παιδιά ώστε κάθε παιδί σε κατάσταση ένδυα να έχει πρόσβαση σε ελεύθερη φροντίδα, ε, στέγαση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη και κατάλληλη διατροφή. Έχει στόχο η Κομισιόν να υποστηρίξει την προσπάθειά μα και μαζί με τα κράτη-μέλη να δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο και ένα σύστημα για να αναπτύξει ένα τέτοιο είδο εγγύηση για τα παιδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ναι, η, παιδιά, η παιδική ένδυα μεταξύ των παιδιών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, λέει η κυρία Τάισεν. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες και είναι οι κυρίως θυγόμενες αυτή τη στιγμή οι οικογένειες αυτές. Το πρόβλημα μεταφέρεται από την πιο ηλικιωμένη γενιά στην πιο νέα γενιά και ιδίως αυτούς που έχουν νέα παιδιά. Εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες των καθόλου μελών για μια μεγαλύτερη κοινωνική προστασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής από την αρχή λοιπόν να έχουμε υπηρεσίες για τις οικογένειες ώστε τα παιδιά να μην είναι οι μεγάλοι χαμένοι όταν οι γονείς τους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή δυσκολίες απασχόλησης. Αυτό λαμβάνει υπόψη στις αναχώρα <clears throat> συστάσεις. Οι αναλύσεις μας λαμβάνουν υπόψη λοιπόν το στοιχείο της ένδυας. Η πολιτική λοιπόν λαμβάνει υποψη λοιπον το στοιχειο της κοινωνικής ενεργοποιηση της κοινωνικης προστασιας θα πρέπει <clears throat> να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να ενισχύσει τις ικανότητες των εργαζομένων ή μη εργαζομένων και να του επιτρέψει να βρουν μια θέση εργασία. Ο καλύτερος τρόπος για να βγει κανεί από την ένδια είναι να βρει μια θέση εργασία. Το να υπάρξει τώρα ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για να εγγυηθεί την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρατε εσεί. Δεν έχουμε ακόμα κάτι τέτοιο. Πρέπει φυσικά να σκεφτούμε σε ποιο μακροπρόθεσμο επίπεδο στο να έχουμε ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Ταμείο το οποίο θα λειτουργεί ως αυτόματος σταθεροποιητής αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν τα μέσα για να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη δεν μπορούμε λοιπόν αμέσως να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα αλλά σε πιο μακροχρόνιο επίπεδο αυτή η ελπίδα μπορεί να υλοποιηθεί αλλά πρέπει να κάνουμε τι απαραίτητε πολιτικέ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τι οικογένειε οι οποίε έχουν νέα παιδιά, γιατί αυτό είναι τμήμα τη κοινωνική μα πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα ερώτημα προς την κυρία Τάισεν. Πρώτα απ' όλα, κάνατε αυτή τη διαπίστωση που είναι πολύ σημαντική ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κοινωνικοί εταίροι. Δεύτερον, η εμπροστοφόρτηση που θα πρέπει να έχει προδραστικό χαρακτήρα και εδώ καταλαβαίνω ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημοσιεύσετε μέχρι το τέλος του χρόνου την κατάσταση των κρατών τι ακριβώς έχουν κάνει με τα χρήματα αυτά για την δημιουργία δομών αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Προς τον κύριο Αντιπρόεδρο, διορθώστε με αν θέλετε οι κατάλληλες αποδοχές, τα δικαιώματα των εργαζομένων, ο ελάχιστος μισθός, χωρίς καμία ε, κάπως ε, κάποια ομαλοποίηση και εναρμόνιση της ε, πολιτικής στα κοινωνικά θέματα. Αυτή είναι η γραμμή που ακολουθεί η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριος Δομπρόφσκης. Εντάξει. Για το θέμα του ελάχιστου, των ελάχιστων αποδοχών. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές εδώ το θέμα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προωθήσει τις συζητήσει και με τα κράτη-μέλη, να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε σταδιακό επίπεδο και να εισαγάγουν ένα επίσημο κατώτατο μισθό στις χώρες αυτές που δεν έχουν κάτι τέτοιο και να εξασφαλίσουμε ότι οι μισθολογικές αυξήσεις συνάδουν με την αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι σαφής λοιπόν η πολιτική μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την κοινωνική πολιτική, δεν θα έλεγα ότι θέλουμε να έχουμε εναρμόνιση της κοινωνικής πολιτικής, γιατί η κοινωνική πολιτική εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχει πολύ περιθώριο όμως για περαιτέρω συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών και αντιμετώπιση με διαμεθοριακών πτυχών της κοινωνικής πολιτικής που μας ενδιαφέρει τα μάλλα. Ευχαριστώ. Δεν μπορείτε να, να θέτε ερωτήματα και στους δύο επιτρόπους, η κυρία Τέισεν η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν που αναφέρεται για την απασχόληση των νέων. Θα προκύψει μια έκθεση και η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς θα εγγύψουμε και στα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης. Τα κρατημέλη θα πρέπει να δώσουν ενδείξεις επί τη βάση μιας σειράς δικτών. Θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και θα τα αναλύσουμε. Κυρία Τρεβέσιους δύο ερωτήσεις προς την κυρία Τάισεν. Μιλήσατε για την χρηματοδότηση προς την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και τα μέσα, τα μέτρα τα οποία θέλετε να αναλάβετε. Θα σας ρωτήσω τι προβλέπετε να κάνετε για να υπάρξουν ελεκτικοί μηχανισμοί ώστε να ελέγξετε ότι αυτή η πρωτοβουλία των νέων πράγματι θα έχει αποδοτικό χαρακτήρα, θα είναι αποτελεσματική. Έχουμε μια ανεργία πάνω του 50% στην Ελλάδα και εκεί είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, σαν παράδειγμα. Επίσης θέλετε να έχετε περισσότερη χρηματοδότηση για τις ε, θέσεις ε, που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, αλλά έχουν ήδη περικοπεί κονδύλια τα οποία συνδέονται με την έρευνα. Θα υπάρξουν λοιπόν τα απαραίτητα κονδύλια, θα επιστραφούν τα απαραίτητα κονδύλια στον τομέα της έρευνας κυρία Τάισεν. Τι θα κάνουμε για να ελέγξουμε την χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για τους νέους. Έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας όταν η Ευρώπη δαπανά κονδύλια υπάρχει ένας δημοσιονομικός έλεγχος ο οποίος ασκείται στην εκταμίευση των κονδυλίων αυτών. Και για τους ποσοτικούς δείκτες. Δεν περιοριζόμαστε σε αυτούς, θέλουμε και να υπάρξουν και ποιοτικά στοιχεία για την πρωτοβουλία των απασχόλησης των νέων. Έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες λοιπόν για τα θέματα αυτά και τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι υπερβολικά αυστηροί οι κανόνες μας αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σωστή χρηματοδότηση των κονδυλίων και θα πρέπει να είναι ποιοτικά θετικό το στοιχείο αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, βασική εκπαίδευση και για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό σε διάφορα επίπεδα. Ξέρουμε ότι 20% των πολιτών μας έχουν ουσιαστικά περιορισμένες ε, ικανότητες σε επίπεδο ανάγνωσης και αριθμητική. στάτομα αυτά λοιπόν δεν έχουν τι απαραίτητε βασικέ ικανότητε για να βρουν μια θέση εργασία και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Κύριο Μπάλα. Όπως είπε και η κυρία Στάινρουκ, έχουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων ε, και πρέπει να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και για την ελευθερία της μετακίνησης, όχι μόνο να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίσεις των επιχειρήσεων, αλλά και των υπαλλήλων. Ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι υποτίμησε τον αντίκτυπο της λιτότητας στην Ελλάδα γιατί είπαν ότι έκαναν λάθος σε κάποιες αξιολογήσεις ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα ε, και το ερώτημα που έχω να σας κάνω είναι το εξής. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είναι το εργαλείο συντονισμού των, πολιτικών, των οικονομικών πολιτικών σήμερα έχετε τα μέσα να δείτε τον αντίκτοπο των ειδικών αναχώρα συστάσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή υπάρχει μία μελέτη ή κάποιες μελέτες που να μπορούν να δουν το μακροοικονομικό αντίκτυπο των ετοιμάτων που ε, έχετε αναχώρα γιατί διαφορετικά μπορεί να προβούμε σε σφάλματα πολύ σοβαρά. Υποθέτω ότι είναι προς τον κύριο αυτή η ερώτηση έχετε το λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές ε, και για τις ειδικέ αναχώρας συστάσεις και για ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Βεβαίως, ε, όταν δημοσιεύουμε τέτοιου είδους συστάσεις, βασιζόμαστε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει της, έρευνας, της ανάπτυξη έρευνας ανάπτυξης για την ενίσχυση της επένδυσης, για την εστίαση στις διαστατικές αλλαγές, όπως επίσης και στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και όλες αυτές τις προτεραιότητες τις μεταγράφουμε σε συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής για τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως όταν προετοιμάζουμε τις ειδικές αναχώρασεις τάσεις, αξιολογούμε το πώς αυτές οι συστάσεις θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη και τις προοπτικές ε, ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε ε, κάθε κράτος Οπότε πρώτα υπάρχουν εκθέσεις που αξιολογούν τις οικονομικές προκλήσεις και στη συνέχεια ακούμε προτάσεις, σχόλια από ε, τους κοινωνικούς εταίρους στα κράτη-μέλη και δεδομένων των προετήτων που ανέφερα προηγουμένως ε, και βάσει των σχολείων που λαμβάνουμε από τις χώρες ε, εκδίδουμε συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η κυρία Σοντέρ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα μου είναι προς την ε, κυρία Τάισεν. Για την κινητικότητα θα ήθελα να ρωτήσω. Ε, σημείωσα τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν, όπως επίσης και ε, τις ε, πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την κινητικότητα. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω να πω ότι η κινητικότητα πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τους νέους. Όμω θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια εμπόδια που υπάρχουν σήμερα, που παρεμποδίζουν αυτή την κινητικότητα σε κάποιες χώρες ε, και ειδικότερα στις διαμεθοριακές περιοχές, όπως αυτή που προέρχομαι εγώ, κάποιοι εταίροι ε, προσπαθούν ακριβώς ε, να βοηθήσουν τον κόσμο να περάσει από το, τη μία χώρα στη γειτονική χώρα. Για παράδειγμα, αυτοί οι φορείς είναι το ε, το διαμεθοριακό ε, ρες, το οποίο είναι πάρα πολύ δυναμικό, ε, είναι πολύ ενθουσιώδης στην ανάληψη δράσης τους, αλλά είναι και πολύ αποθαρρυμένη από το άχθος που υπάρχει όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη ακριβώς προς όφελος της δράσης ενίσχυσης της κινητικότητας. Εκεί στο παρελθόν είχαμε τρία χρόνια ε, τριετή προγράμματα, τώρα έχουμε μονοετή προγράμματα, οπότε έχω την εντύπωση ότι αποθαρρύνονται αυτοί οι φορείς που διευκολύνουν την κινητικότητα. Δεύτερον, εκμάθηση γλωσσών. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημά Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Προτάσεις θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν ε, για την εκμάθηση των γλωσσών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας, ε, κυρία ε, Σοντέχ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά του ΡΕΣ και Υπάρχουν κανόνες που διαδιευκολύνουν ε, τη ζωή των ανθρώπων που πρέπει να το εφαρμόσουν. Ε, για το οικονομικό κομμάτι η κυρία ε, Γεωργίεβα το γνωρίζει αυτό και προσπαθεί να δει πώς μπορεί να απλουστευτεί η κατάσταση, οι οικονομικοί κανόνες που επίσης θα βοηθήσουν την ε, ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών. Όσον αφορά τη κινητικότητα και το διαμεθοριακό χαρακτήρα, δεν θέλουμε μόνο να ενισχύσουμε το ΡΕΣ και είναι κάτι που έχει αρχίσει ήδη. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του δικτύου των υπηρεσιών απασχόλησης των διαφόρων κρατών μελών. Προσπαθούμε να τους συντονίσουμε, να συνεργαστούν και ακούω ε, ότι επί τόπου δουλεύει αυτό και είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει βεβαίως και να βελτιώσει τη ΡΕΣ γενικότερα. Ο κύριος Σάιμον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, Μήπως μπορείτε να μας πείτε για, τους αποσπα... για την απόσπαση των εργαζομένων. Μπορείτε να μας δώσετε μια σαφή απάντηση. Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τη συγκεκριμένο κανονισμό, δεν νομίζω ότι επαρκεί αυτό που μας είπατε. Ε, πρόκειται εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουμε δημοψήφισμα για το αν θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασική ερώτηση είναι για ποιο λόγο έρχονται ξένοι εργαζόμενοι ε, εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο να δουλεύουν και μειώνονται οι μισθοί δικοί μας ε, ε, υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι προστατεύονται από την οδηγία για την απόσπαση. Ε, ε εσείς ως ε, Επίτροπος, πρέπει να το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μια νέα οδηγία απόσπασης που πραγματικά θα προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς και όταν ε, μας ζητούσε υποστήριξη για να εκλεγεί ο κύριος Γιούγκερ μας το υποσχέθηκε αυτό. Κάτι που θα κάνει δίκαιη την αγορά εργασίας και που θα κρατήσει ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τεράστιες διαφορές. Αν δεν το λύσετε αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι η τελευταία χώρα που θα φύγει. Ευχαριστώ πολύ είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην συγχαίουμε την ελευθερία μετακίνησης με την απόσπαση των εργαζομένων. Διότι πρώτα απ' όλα η ελευθερία της μετακίνησης ε, είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου και ο πρόεδρος κύριος Γιούγκα ε, είπε ότι οι τέσσερις ελευθερίες ε, δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν τη βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το θέμα της απόσπασης εργαζομένων είναι πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αφορά κάποιες εταιρείες όπου ε, αποσπώνται εργαζόμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε μια άλλη χώρα. Υπάρχει αυτό το θέμα στην οδηγία και όταν ανέλαβε η καινούργια επιτροπή πράγματι δεσμεύτηκε ε, στο ότι θα αναθεωρητήσει αυτή την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Αυτό κάνουμε τώρα με την Επίτροπο κυρία Τάισεν, δηλαδή δουλεύουμε πάνω σε αυτή την οδηγία, αλλά σας λέω και πάλι αυτό δεν θα πρέπει να το συγχαίρετε με την ελευθερία μετακίνησης. Ο κύριος Ρολόν. Κύριε Επίτροπε, θέλω να επανέλθω στο θέμα του κοινωνικού διαλόγου. Αναφερθήκατε στο θέμα αυτό και συμφωνώ μαζί σας. Είναι καταρχήν θέμα των κοινωνικών εταίρων ο κοινωνικό διάλογο, αλλά η Κομισιόν <clears throat> έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Έχει μια μεγάλη ευθύνη να επομιστεί το να δημιουργήσει το πλαίσιο που θα επιτρέψει τον κοινωνικό διάλογο και να εξασφαλίσει ότι αυτό ο διάλογο δεν είναι μονάχα μια ρητορική ανταλλαγή απόψεων, αλλά οδηγεί σε συγκεκριμένε συμφωνίε, οι οποίε στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμοστούν και τονίζω σχετικά τη Συμφωνία των Αυτονόμων Συμφωνιών. Έλαβε χώρα μια συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου, τώρα οι κοινωνικοί εταίροι προσπαθούν να τελειώσουν το έργο τους για τα προγράμματα. Υπάρχει η κατάλληλη όθηση λοιπόν και ορμή για να μπορέσουμε να, να ε, επαναεκκινήσουμε τον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ, κοινωνικό, πολύ σημαντικός. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μια πιο εύκολη πτυχή για τους κοινωνικούς εταίρους για να προχωρήσουν όπου υπάρχει μια ανάλυση στα θέματα της μαθητείας, της κατάρτισης, της εναλλαγής. Αν μπορούμε εκεί πέρα να τους παρατρύνουμε να συμφωνήσουν σε κάτι, να έχουν μια συμφωνία που θα ενισχύσουν την δική μας ε, ευρωπαϊκή πολιτική για την εναλλακτική, για την κατεναλλαγή μάλλον μαθητεία και για να αντιμετωπίσουμε έτσι και την έλλειψη θέσεων εργασία. Καλά λέει ο κύριος Σταμπρόφσκης για τον κοινωνικό διάλογο. Είναι φανερό, όπως είπαμε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και το έχει πράξει ήδη στο παρελθόν με το να ενισχύσει και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πιο πρόσφατα με το να δώσει ειδική μνήμα στο ρόλο των αυτονόμων συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων μέσα στο πλαίσιο της καλύτερης νομοθεσίας Τώρα υπάρχουν εξαιρέσει σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες εκθέσεις αντικτύπου και τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό καθεστώς των κοινωνικών εταίρων όπως αναφέρονται στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίδων στις αυτόνομες συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων ένα διαφορετικό είδος μεταχείρισης από ό,τι έχουμε στην Γενική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει ότι έχει ένα ρόλο διευκολυντή και του διμερούς διαλόγου ώστε να μπορέσει να επιτύχουν οι κοινωνικοί εταιροί αυτές τις ε, αυτόνομες συμφωνίες αλλά αυτό πάντα μπορεί να το κάνει στο τέλος της ημέρας η Κομισιόν όταν μιλάμε για τον διημερή αυτό διάλογο είναι μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων το να συμφωνήσουν. Μπορεί να συμμετάσχει λοιπόν και η Κομισιόν σε ένα τριμερή διάλογο και ε, διερευνούμε νέους τρόπους να συμμετάσχουμε και να ενισχύσουμε τους κοινωνικούς εταίρους και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαβουλεύσεις με αυτούς. Ευχαριστώ, κ. Ευχαριστώ, ο Μέσω της ε, Προέδρου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο και την κυρία Τάισεν για το γεγονό ότι ήρθαν εδώ για να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Άκουσα στην απάντησή σα στη συνάδελφο από την Ιταλία ότι παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην Ιταλία και ερωτώ παρακολουθείτε και τις εξελίξεις μήπως στη Βρετανία, στη δική μου τη χώρα, γιατί είναι ένα λαμπρό παράδειγμα επιτυχίες, η πιο επιτυχημένη οικονομία στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Έχουμε από το 2010 άλλες 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και πρόκειται να ε, θεσπίσουμε, να ε, κατασκευάσουμε άλλες, ε, άλλα δύο εκατομμύρια θέσει απασχόλησης. Άρα δηλαδή όλοι θα έχουν θέση εργασίας και πώς το κάναμε αυτό με το να καταστεί απασχόληση πιο ελκυστική από την απέλπιδα ανεργία. Η πρόνοια δεν είναι επιλογή. Βεβαίως Εκείνο το οποίο καταφέραμε είναι να ρυθμίσουμε τα φορολογικά. Όποιος βρίσκεται με ελάχιστο μισθό στη χώρα μου ε, δεν πληρώνει φόρους ή περίπου. Έγινε λόγος για την ανεργία των νέων. Τα πανεπιστήμια είπατε ότι είναι ένας ε, τρόπος για να εξοικειωθούν οι άνθρωποι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να σας πω ότι και η μαθητεία είναι η απάντηση. Εμείς στη Βρετανία είμαστε δεσμευμένοι να προσφέρουμε 3 εκατομμύρια θέσεις μαθητείας και ε, ρωτώ γιατί δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες θέσεις μαθητείας στην Ευρώπη προσφέροντας τους ε, εργοδότες, τους εργαζόμενους που πραγματικά χρειάζονται. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κυρία Τάισε, νομίζω η ε, ερώτηση τέτοι προς εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εμείς ε, στην Ευρώπη προσπαθούμε να προάγουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές τα κράτη-μέλη μπορούν βέβαια το ένα να μάθουν από το άλλο για να αποφύγουν δυσκολίες. Όσον αφορά τις θέσεις μαθητείας, εμείς ζητάμε από τους εργοδότες να εγγυώνται τις θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα πάλι στις θέσεις μαθητείας, προσπαθούμε να δούμε πώς είναι δυνατόν να είναι πιο φυσιολογική η μαθητεία, δηλαδή τι μορφή μαθητείας μπορούμε να προσφέρουμε και η κατάσταση ποικίλει από μέλος σε μέλος, από κράτος σε κράτος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα κάνω μια ε, πολύ, ε, δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, λέει κυρία Ραντκε. Θέλω να γνωρίζω εσείς τι πιστεύετε σχετικά με τις ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές που χρειαζόμαστε πηγόντως αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσείς προτίθεστε ε, να προτείνετε ε, μια ελάχιστη κοινωνική προστασία σε αυτά τα, ε, τις νομοθετικές πράξεις, πράξεις που θα καταθέσετε. Πράγματι έχουμε ένα κοινωνικό θεματολόγιο, λέει η Επίτροπος, και μας ενδιαφέρει να εμβαθύνουμε ε, γενικότερα στα ε, κοινωνικά προγράμματα. Αν τώρα με ρωτήσετε για την προσωπική μου θέση, στην τελική ανάλυση αυτό που μετράει είναι περισσότερο η θέση του κολεγίου. Προφανώς και συζητάμε οι επίτροποι ανάμεσά μας, αλλά αυτό που μετράει είναι η θέση του σώματος των επιτρόπων. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με το να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές ε, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας για να μην υπάρχει αυτή η καθοδική περιδίνη Πάντω Πάντως οι ε, αρμοδιότητές μας, ε, όπως είπε και ο κύριος Ντομπρόφσκι, πολλές φορές επικαλύπτονται με αυτές των κρατών μελών. Εάν λοιπόν τα κράτη-μέλη θέλουν να καλύψουν αυτό το στόχο, τότε πράγματι πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν και δείκτες για την ελάχιστη κοινωνική ε, προστασία. Αυτό ισχύει και για το ελάχιστο εισόδημα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και στους δύο επιτρόπους που είναι παρόντες εδώ. Πάρα πολύ απλά ερωτήματα σε σχέση με τις, τα επιδόματα ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν το έχει εγγράψει στην μέση διαταξή της το είχε εξετάσει με τους αρμόδιους υπουργούς και έχει ε, κάνει και μία έκθεση, η Κομισιόν έχει επιφορτήσει τη δημιουργία μιας μελέτης για τα τεχνικά θέματα για το ζήτημα αυτό. Με ενδιαφέρει και η κοινωνική διάσταση και η ανάγκη να διευρύνουμε τον κοινωνικό τομέα στην περιοχή του ευρώ, αλλά και τα μακροοικονομικά ζητήματα τα οποία τίθενται. Δεν εμπλέκεται μόνο το θέμα της αλληλεγγύης, αλλά και ο μακροοικονομικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσουμε τους ασυμμετρικούς κλειδονισμούς όπως αυτούς που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν να μου απαντήσει. Uh, okay. Uh, this is... Uh, ναι, αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί μέσα σε ένα πλαίσιο της εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μια εγγύηση για τα επιδόματα ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στις ε, εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, οι πέντε πρόεδροι εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας νέας έκθεσης σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ενώσεως και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους προς το Συμβούλιο των, τους επόμενους μήνες. <clears throat> Δεν μπορώ να προκαταλάβω λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης των πέντε προέδρων, αλλά σε γενικές γραμμές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση οι προτάσεις στο να αντιμετωπίσουν και βραχυχρόνια προβλήματα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα μέσα στην τρέχουσα συνθήκη και πιο μακρο, μακρόπνοα ζητήματα και αυτό που αναφέρατε είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ήταν υποσυζήτηση και στο πλαίσιο της λεγόμενης δημοσιονομικής ικανότητας της ε, ζώνης του ευρώ. Προς το παρόν όμως δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω σε σχέση με το περιεχόμενο της έκθεσης των πέντε πρόεδρων μέχρι ότου οι πέντε πρόεδροι περατώσουν το έργο τους αλλά σίγουρα το θέμα αυτό βρίσκεται στην ε, είναι συνέντευξη των θεμάτων που τους απασχολούν. Παρακαλώ. Η, ο διαρθρωμένος αυτός διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός και ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Προς την κυρία Τάισεν, εγώ είμαι πεπισμένη ότι μία εγγύηση για την απασχόληση θα ήταν ένα πολύ καλό στοιχείο μαζί με τις επενδύσεις στα κράτη-μέλη με την ε, μείωση της ανεργίας μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα όπως στην περίπτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας. Έχουμε όμως προβλήματα με την απασχόληση ε, ατόμων που είναι φτωχά και ζουν στις λεγόμενες αποκλεισμένες περιοχές, σε περιοχές που είναι υποβαθμισμένες. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία για τα θέματα αυτά, ώστε ένα τμήμα του Ταμείου να ασχοληθεί με τα άτομα σε απομεμακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην απασχόληση. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν έχει πολύ περιορισμένε δυνατότητε δράση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη διαδικασία ανοιχτού συντονισμού. Τι μπορεί να κάνει όμως η Κομισιόν είναι καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερη εποπτεία της κατάστασης. Είναι ανεπαρκή τα στοιχεία της Eurostat. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Προβλέπει η Κομισιόν να προχωρήσει σε καλύτερο μηχανισμό εποπτεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το Ταμείο για την Απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για κάποιε ομάδε ε, στόχο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πιο ευάλωτε ομάδε στην κοινωνία μα και πρέπει να μα απασχολήσει αυτό όλο ιδιαίτερω και αυτό κάνουμε στις ε, εκθέσεις ε, και στις συστάσεις αναχώρα. Μπορείτε εκεί να διαπιστώσετε ότι για μερικά κρατημέλη ζητούμε περισσότερη προσοχή σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Υπάρχουν βέβαια διαφορές μεταξύ των χωρών. Η απλοποίηση της χρήσης ε, για ε, την αποδέσμευση των ε, κονδυλίων από τα ταμεία σε ένα πιέσιο πολιετές αποτελεί μια μέθοδο απλοποιημένη. Αλλά πρέπει τα κράτη-μέλη να αποδεχθούν αυτές τις αλλαγές. Όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, ζητήσαμε από τη Eurostat, επειδή χρειαζόμαστε δεδομένα για την αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα κρατη ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη, όπως είπα, να ε, βοηθήσουν λιγάκι, να βιαστούν για να έχουμε πιο νωρίς διαθέσιμα τα στοιχεία και να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρτέν, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας άκουσα και τους δύο πολύ προσεκτικά και Πρέπει να πω το εξή. Ανεργία νέων, των νεότερων, των μεγαλύτερων, εξαφάνιση θέσεων απασχόληση, δημιουργία θέσεων απασχόληση, μείωση τη αγοραστική ικανότητα, ε, ε, βελτιώσει αργά αλλά σταθερά. Αυτό που άκουσα είναι ότι είναι ευσεβής πόθη, θέλουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα ενώ γνωρίζουμε τις αιτίε. Παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση και αυτό το παγκοσμιοποιημένο πρόγραμμα, οικονομικοποίηση της οικονομίας, μεταναστευτικές ροές, οποίες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, δεν μπορούμε πια να τις διαχειριστούμε. Μείωση του σχολικού επίπεδου, λες και θέλουμε να ε, είναι λιγότερο ικανοί οι νέοι για ποιο λόγο δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε επιτέλους τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων. Η κυρία Τάισεν. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την ανάλυση σας. Λέτε ότι δεν, δεν ε, ε, αντιμετωπίζουμε τις αιτίες μεταλλάσσεται η κοινωνία μας. Βλέπουμε την εξέλιξη, εξέλιξη της τεχνολογίας. Υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις, κάτι το οποίο βέβαια δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες. Όμως το να λέμε ότι θα σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση, ε, τι να σας πω, δεν και λύση αυτό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προκλή, κάποιες προκλήσεις, ε, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μία μάχη, όμως γι' αυτό το λόγο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν και πράγματα που τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τα κάνουν μόνα τους. Είμαστε πιο ισχυροί ενωμένοι. Έχουμε συγκεκριμένες αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να ε, απολαύσουμε αυτές τις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να το κάνουμε αυτό και σε επίπεδο εργασίας. Πρέπει να έχουν οι πολίτες επαρκείς δεξιότητες για να μπορούν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα και για τις χώρες τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Όλοι όσοι είχατε εγγραφεί είχατε τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους. Ήσασταν πάρα πάρα πολύ καλοί στις απαντήσεις σας, γρήγοροι. Θα σας προσκαλέσουμε σύντομα ξανά. Γιατί θα έχουμε νέες ερωτήσεις να σας θέσουμε. Τώρα λοιπόν να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Δύο λεπτά να τεντωθούμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τα σωστά χαρτιά μπροστά μας και θα αρχίσουμε σε δύο λεπτά την ψηφοφορία. Λοιπόν, έχετε φαντάζομαι έτοιμες ε, τις ε, προσωπικές σας ε, κάρτες για να ψηφίσετε. Θα προχωρήσουμε. Προχωράμε λοιπόν με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά ψηφορία για την αποτελεσματικότητα των πόρων βαντίζουμε προς μια κυκλική οικονομία. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης ε, και τροπολογίες. Αν λοιπόν είσαστε έτοιμοι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ, τα αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική A, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10. Είναι η 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η B υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται Ισί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική D παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 31. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω, μάλλον μπορεί και να απορρίφθηκε. Καλύτερα εδώ να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πάμε στην... Ψηφίζουμε για την 32 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 υπέρ κατά απορρίπτεται η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ή e, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η G η συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά... Ο, καταπίπτη. συγγνώμη καταπίπτη, λέει η πρόεδρος. Πάμε στην 7, τροπολογία υπαριθμών 7. Μάλλον όχι, στην 57 υπέρ κατά... Λάθος έκανε η πρόεδρος. Με συγχωρείτε. Για την 7 πρώτα, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 7 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 57 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. η συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πενήντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εξήντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 61 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, όχι καταπίπτει, η 67 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης, ως τροποποιήθηκε, ψηφίζουμε παρακαλώ. And the vote is closed. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Uh, Πηγαίνουμε τώρα στο σημείο 11 για την ε, επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Τροπολογία 1, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριπτε. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 εκπίπτει, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Μα πρέπει να ψηφίσουμε τη 14. Αλλά είναι κρίση 13. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα λάθος, έκανα λάθος. Ξαναψηφίζουμε τη 15 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16. Ε, έλεγχος για 15, άρχιε η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται, 16, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική συγκ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 και 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτές 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 31 έλεγχος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 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ή e, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 47 εκπίπτει, συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές Εποχές, πρέπει να ελέγξουμε την 55 55 άρχεται η ψυχοφορία. πέρας απορρίπτεται. το σχέδιο γραμματότης όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση ψηφίσμα ακόμα το σύνολο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Εγκρίνεται. Ωραία. Συνεισφορά της Επιτροπής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 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απολύτω. Τροπολογία 7 έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τροπολογία εννέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ανοίγει περαιτέρω, αλλά τώρα έκλεισε. Εγκρίνεται. Ναι, ναι, πρέπει να ελέγχουμε καμιά φορά. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 εκπίπτει. Τροπολογία 12 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη έλεγχος τροπολογία 13 τμήμα 1 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά Α, εκπίπτει η τροπολογία 14. Πάμε στην τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έργος, για 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη και λιγότερη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος στην 20. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 εκπίπτει. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για 24 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 25, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Θα δούμε σε τελική ανάλυση και σε τελική θεώρηση τι θα γίνει. Κάποιος δεν ψήφισε, πέρα τις προφορίες, εγκρίνεται. Τροπολογία 28, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Ε, ελέγχουμε την 28. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Έχουμε μια συμφωνία για αυτή την προφορική τροπολογία. Θέλω να διαγράψω τη λέξη οδηγία και αντί για οδηγία προτείνω τη λέξη μέτρα. Η οδηγία να γίνει μέτρα. Υπάρχει αντίρρηση. Ψηφίζουμε την τροπολογία 30. με την προφορική τροπολογία. Κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος 31, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 Ελέγχουμε την 32. Πέρας. Απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχος για 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. έλεγχο στην 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει και απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ε, προφανώς. Είναι 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει σιγά σιγά. Έκλεισε. Απορρίφθηκε. Και τώρα η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση για τη συμβολή της Επιτροπής Απασχόλησης για το διαρθρωμένο διάλογο. Άρχεται η ψηφοφορία. Αλλά κλείνει και στη συνέχεια. 37-8 με 0 αποχές. Όχι, άλλη μία, όχι. Αυτό ήτανε. Στις δύο ξαναρχίζουμε. Και κάποιοι από εμάς είναι ευτυχισμένοι. για να προλάβουμε τις πτήσεις μας και τα τρένα μας. Αλλά γυρίστε σας παρακαλώ, να μείνουμε μόνοι μου γιατί νιώθω μοναξιά. Σας ευχαριστώ.